Ανανεώνεται τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πρακτικά της χθεσινή ε, συνεδρίασης και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Έχετε αντιρρήσεις σχετικά. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά λοιπόν.